Right, welcome back everybody. I... Καλημέρα. Καλώς ήρθατε μετά τις διακοπές. Ελπίζω να περάσατε ωραία. Ζητώ συγγνώμη από τώρα. Αν με δείτε να εξαφανίζομαι κάποια στιγμή, να ξέρετε ότι έχω ένα πρόβλημα με την πλάτη μου και δεν μπορώ να κάθομαι συνέχεια. Δεν έχει λυθεί ακόμα το πρόβλημα αυτό με το σωστό εξοπλισμό, τις σωστές καρέκλες εδώ. Οπότε να ξέρετε ότι θα είναι γι' αυτό. Το πρώτο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι ως ήθιστε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Επίσης θέλω να σας υπογραμμίσω εδώ ότι τα σημεία 3 και 4 που είναι για μια αυθεντική οικονομική και νομισματική ένωση που συζητάμε και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Τράκη και που με τον κύριο Μπαρνιέ θα έχουμε επίσης ανταλλαγή απόψεων, θα γίνει και κλεισμένον των θυρών η συζήτηση αυτή. Και ο λόγος είναι για να μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία ίσως δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν ακόμα. Άρα τα μέσα ενημέρωσης ότι λόμπι βρίσκονται εδώ θα πρέπει να βγουν από την αίθουσα για ε, το σημείο αυτό. Εννοείται ότι οι άνθρωποι του Κοινοβουλίου μπορούν να μείνουν οι ευρωβουλευτέ και αυτή τη Επιτροπή αλλά και άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, γιατί υποθέτω ότι θα έρθουν και ευρωβουλευτέ από άλλε επιτροπέ που θα θέλουν να παρακολουθήσουν και οι βοηθοί μπορούν να παραμείνουν στην αίθουσα τότε. Αλλά όποιο δεν είναι προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να βγει από την αίθουσα τότε και στις 6.30 ε, μετά θα συζητήσουμε άλλα πράγματα με τον Όλυ Ρεν που έχουν να κάνουν ε, με το ευρώ κλπ. Οι υπόλοιπε ανακοινώσεις θα γίνουν στις 5.30. Συνεπώς, περνάμε τώρα στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης που είναι η δυνατότητα εισαγωγής των ομολόγων σταθερότητας. Και δίνω τον λόγο στην εισηγήτρια, την Σιλβή. Ευχαριστώ πολύ Σάρων. Λυπάμαι για σένα, για την πλάτη σου δηλαδή, αλλά εγώ χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ. Λοιπόν, δεν θέλω να χάσω πολύ χρόνο. Ευχαριστώ τους ναδέφους για τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει και που είναι πολλές. Αυτό πάντως που θέλω να κάνω τώρα είναι να ακούσω πρώτα τους συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες. Έχουμε ήδη συνεργαστεί με τους σκιώδεις, οπότε ξέρουμε λίγο πολύ τις θέσεις των διαφόρων ομάδων. Κατά τα άλλα υπάρχουν πράγματα που είναι σε εκκρεμότητα, όπως είναι το θέμα του μηχανισμού σταθερότητας. Οπότε αν συμφωνείτε να αρχίσει η συζήτηση, να ακούσω έτσι ποια είναι η γενική αίσθηση στην αίθουσα και μετά να πάρω το λόγο παρακαλώ. Καλώς λέει η Πρόεδρος, ήσουν πολύ γρήγορη, πολύ σύντομη. Παρακαλώ, κύριε Θεό, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σάρων και θέλω να ευχαριστήσω και να χαιρετήσω όλους τους συναδέρφους που ήρθαν εδώ για αυτή την πρώτη ε, συνεδρίασή μας. Θα είμαι και εγώ σύντομος. Τώρα θα αρχίσουμε την συζήτηση επί των τροπολογιών. Ως σκιώδης συζητητής προσπάθησα να υποβάλω τροπολογίες που να βρίσκουν σύμφωνους όλους στο ΕΛΚ οι δυνατόν. Όπως επίσης προσπάθησα να υποβάλω και τροπολογίες με τις οποίες να συμφωνούν όλοι στην αίθουσα εδώ. Να ξέρετε ότι οι τροπολογίες μου ακολουθούν δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι το ταμείο εξόφληση, δηλαδή πώς θα βάλουμε μαζί το χρέος για να εξοφληθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πανάκια βέβαια, ότι πρόκειται για ένα θαύμα, ότι θα γίνει εξυγίαση ευθύ αμέσω. Δεν είναι κάτι που βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πετύχουμε. Μέσο πρόθεσμα όμω. Μεσοπρόθεσμα ναι. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για το μέλλον. Αυτό, είναι... Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις συνθήκες και να έχουμε μια ενισχυμένη οικονομική ένωση με μια κυριαρχία στον προπολογισμό και έναν σταθερό μηχανισμό προπολογισμού. Είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μία λύση με δημοσιονομική πειθαρχία σε επίπεδο όλων των χωρών μελών. Έτσι λοιπόν με τις τροπολογίες μου προσπαθώ να συνεχίσω με την ιδέα του χαρτιπορίας που προτείνει και η συγκήτρια. Και εγώ ίδιος κάνω μια πρόθεση, μια πρόταση, συγγνώμη, ε, βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη, με τα European Safe Bonds, δηλαδή για τα ευρωπαϊκά αποταμιευτικά ομόλογα. Αυτά δεν είναι ακριβώς ε, μια κοινή εγγύηση, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια πρόταση η οποία αξίζει να μελετηθεί πιστεύω σε βάθος. Κατά τα άλλα, μακροπρόθεσμα δηλαδή, πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μηχανισμούς αποτελεσματικούς εποπτείας των προπολογισμών με ένα πραγματικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τροποποίησεις ενδεχομένως στις συνθήκες μεγάλες. Αυτές είναι οι ιδέες λοιπόν που εγώ έχω να προτείνω. Κατά τα άλλα είμαι στην διάθεσή σας προκειμένου να συνεργαστώ με όλου τους συναδέρφους εδώ αλλά και όλους τους υπόλοιπου για ό,τι θέματα πιστεύετε ότι είναι σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρο Από τους συσσελιστέ είναι εδώ κανεί. Όχι. Κύριε Έπινγκ. Α, ούτε και ο κύριος Έπινγκ είναι εδώ. Φιλίπ, εσύ, η σειρά σου. Ευχαριστώ, Σάρων. Ελπίζω να ευσταθείς καλύτερα σύντομα. Καλώς ήρθατε όλοι πάλι στις Βρυξέλλες. Θα μιλήσω γαλλικά, λέει ο μιλητής, μια που και η συγγήτρια μεγαλόφωνη. Η δουλειά που έκανε είναι μια δουλειά ακροβάτη. Προσπαθεί να πετύχει μια καλή ισορροπία. Έχω μιλήσει και με τον Τιέγο για το θέμα αυτό της ε, αποκοινού διάθεσης και εξόφλησης του χρέους. Είναι κάτι που μπορούμε να πετύχουμε μεσοπρόθεσμα. Θέλω να πω στον Διέγκο ότι ναι, αυτό είναι ένα μέσο, ένας μηχανισμός μόνο, αναγκαίος βέβαια. Και έπειτα ε, ναι μεν μπορεί να πετύχει κάτι μεσοπρόθεσμα, μόνο μεσοπρόθεσμα, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε με το μεσοπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα τι είναι. Εγώ στον ιδιωτικό τομέα ξέρω ότι είναι τρει μήνε. Αν το μεσοπρόθεσμα για μένα είναι 12 μήνε, τότε δεν έχω πρόβλημα. Αν βέβαια είναι 12 χρόνια, τότε έχω πρόβλημα. Γιατί αν θέλουμε να λύσουμε την κρίση, αυτή την κοινή κρίση που έχουμε με τα δημοσιονομικά μας στην Ευρώπη χωρίς αυτό το μηχανισμό. Δηλαδή πρώτα να λύσουμε την κρίση και μετά να δούμε αν θα βάλουμε μαζί το χρέος από κοινού ή όχι. Ερχόμαστε στη συζήτηση αυτών που λένε να έχουμε πρώτα μια πολιτική ένωση, αλλά πρώτα έχουμε μια τραπεζική ένωση και μετά βλέπουμε πώ θα διαχειριστούμε από κοινού το χρέο. Ενώ από την άλλη υπάρχουν αυτοί που λένε όχι, πρώτα να φτιάξουμε την ένωση του Χρέου και μετά να δούμε για την τραπεζική ένωση και την πολιτική ένωση. Μα έχουν άδικο και η μεν και η δε, γιατί αυτά όλα πρέπει να γίνουν μαζί. Δυστυχώ δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε και να καθίσουμε να σκεφτόμαστε άλλα 10 χρόνια. Συνεπώ η δικιά μα η θέση είναι αυτή που λέει. Καταρχήν, ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε όπως λέμε και για τα πυρηνικά. Ακόμα και αν ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνο, την απόφαση πρέπει να την πάρουμε τώρα. Και μετά σιγά σιγά να την θέσουμε σε εφαρμογή. Έπειτα δεν μπορούμε να βάλουμε από κοινού το χρέος και να εξοφλήσουμε από κοινού το χρέος χωρίς συγχρόνως να έχουμε οικονομικές δεσμεύσεις που να έχουν λάβει εκείνοι τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε δημοκρατικά. Συνεπώς, πρώτον, δεν μπορεί να παραμείνει ακαδημαϊκή η συζήτηση, πρέπει στην πράξη να δούμε τι θα κάνουμε και δεύτερον να φροντίσουμε για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή ε, το σύστημα της αποκίνου εξόφλησης του χρέους χωρίς να έχουμε πραγματικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι ε, βάζουμε από κοινού και την κυριαρχία, την κάνουμε συλλογική. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε για αργότερα. Συλλογικά λοιπόν, αλλά και ατομικά, όλες οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν 100% κυριαρχία. Πρόκειται για ένα θέμα συλλογικού ε, συμφέροντος πάντως και όχι ατομικό. Το τρίτο που θέλω να πω είναι το εξή. Μπαίνουμε σε έναν διακυβερνητικό δρόμο δεν θα μάθω την κοινοτική μέθοδο εγώ στη Σιλβή, μάλλον η Σιλβή θα τη μάθει σε μας. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι πολύ βασικό αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, το ιδεώδε δεν είναι να έχουμε έναν επίτροπο για τα οικονομικά και νομισματικά, ο οποίο να δρά μόνο του χωρί έλεγχο και ο οποίο να αντικαθιστά τα κοινοβούλια ή τι εθνικέ κυβερνήσει. Όχι, μια επιτροπή θέλουμε η οποία να λογοδοτεί σε εμά και η οποία να μπορεί να ανακληθεί εφόσον σφάλει στις πολιτικές της εκτιμήσεις. Επίσης γίνεται εδώ πέρα και μία σύνδεση με την σημερινή κατάσταση. Δηλαδή εμείς πιστεύουμε ότι η Κομισιόν δεν αποφελείται την ελαστικότητα που μπορεί να έχει όσον αφορά την μακροοικονομική, το μακροοικονομικό και δημοσιονομικό έλεγχο των χωρών και μερικές φορές ε, το... είναι υπερβολικά αδύναμη. Δηλαδή δεν προστατεύει ούτε καν τις επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στο μεταπηδικό τομέα στις οικονομίες μας. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έδειξε ότι δεν είναι κάτι που είναι πρωταρχικό στη δράση της Κομισιόν. Επίσης δεν είναι πω στον Τιέκο παρόλο που μπορεί να μην τα λέω ακριβώς όπως τα σκέφτεσαι εσύ, ακόμη και αν σήμερα αποφασίσουμε ότι βάζουμε από μαζί την εξόφληση του χρέους, αν θέλουμε να το κάνουμε δημοκρατικά αυτό, χρειάζεται χρόνο. Η δημοκρατία απαιτεί χρόνο. Τι να κάνουμε, είναι φυσιολογικό αυτό. Το μόνο σοβαρό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μα για να αγοράσουμε εντό αγωγικών τον χρόνο που χρειαζόμαστε, είναι να έχουμε αυτή τη μεγάλη μπαζούκα που λέγαμε. Δηλαδή, ο μηχανισμός ευρωπαϊκός σταθερότητας διαθέτει όλα τα μέσα που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Και συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι διακριτή η ρόλη. Δηλαδή, ε, ο Ευρωπαϊκός ο Χρηματοπιστωτικός Μηχανισμός να έχει διακριτό ρόλο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά δεν πρόκειται να το καταφέρουμε αυτό χωρίς να ε, μπορούμε τραπεζικά να το δούμε. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι προτάσεις έρχονται τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά. Ο Σαρκό ήταν ο πρώτος που ήρθε, ο Σαρκοζή μετά ήταν ο Μόντι. Η τραπεζική άδεια για μας, συλλογικά τους Ευρωπαίους, είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για να φτιάξουμε την πολιτική και την τραπεζική ένωση που θέλουμε και την ένωση του χρέους. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να οδηγηθούμε στην κατάρρευση, κάποια μέρα και όσο γίνεται πιο γρήγορα τόσο καλύτερο, να αποφασίσουμε για αυτήν την τραπεζική άδεια το ευρω... στο ΕΜΣ. Υπάρχει κανείς από την ο η συνάδελφος ε, που είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό, αρμόδια, αν θέλετε δεν έχει έρθει ακόμη, θα έρθει αργότερα, γι' αυτό δεν έχω κάτι να πω. Πρόεδρος, έχω δύο μιλητές στον καταλογό μου, υπάρχει κάποιος άλλος, Άστριτ. Uh, Mrs. Trezic, Ivo, anybody else? Άλλος. Wolf. Έχεις το λόγο. Όλοι συμφωνούμε, φαντάζομαι, ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια δύσκολη κατάσταση της οποίας τη λύση δεν μπορούμε να τη βρούμε εμπειρικά. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Η, τα μπλε και τα κόκκινα ευρωομόλογα, μετά τα μπαζούκα, Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Ένωση κλπ. κλπ, κλπ. Έχω πρόβλημα, έχω πρόβλημα και ε, με το έγγραφο, με το σχέδιο εκθέστης της συνάδελφου Γκουλάρ α, για το γεγονός ότι ε, ξεκινούμε μεν με το δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο υποστηρίζω και εγώ και τα λοιπά ναι, αλλά μετά προχωρούμε και μιλάμε για κοινά ομόλογα α, ναι, 25 ετών και λοιπά και λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κοινοτικοποιήσουμε ή εν να αναλάβουμε την αποκοινού εξόφληση του χρέους 100% όλοι μας τα μπλε και τα κόκκινα ομόλογα συν όλα τα άλλα που προτείνονται εδώ οδηγούν σε κατά 100% τα εκατό εξόφληση του χρέους από κοινού. Αυτό το θεωρώ λανθασμένο και από νομική άποψη και από πρακτική άποψη. Ε, ξεχνάμε ε, ότι ότι ε, λέγοντας κάτι τέτοιο είναι σαν να ξεχνάμε και να παραπελμελούμε τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν για αύξηση ανταγωνιστικότητας κλπ. κλπ. Και ανάπτυξη. Δεν... Ε, το προσωπικό μου πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό και βεβαίως δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί Ας ξεκινήσουμε αργά-αργά. Ας ξεκινήσουμε με ένα πρώτο μηχανισμό μαζί με το EFSF και μαζί ίσως και με αυτά που θα μας πει ο κύριος Δράγκη να βάλουμε, να ξεκινήσουμε μια πορεία και βλέπουμε αργότερα τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μαζί στο τραπέζι. Ας περιοριστούμε σε αυτά που θεωρούμε αυτή τη στιγμή σωστά και εφικτά. Ευχαριστώ. Λέων, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια τη Σιλβή που ανέλαβε να ξεκινήσει τον αγώνα αυτό για τα ευρωομόλογα ε, που είναι στόχος των για τη δημιουργία μιας φεντεραλιστικής Ευρώπης και που τον υποστηρίζουμε. Εμείς που πιστεύουμε σε αυτή την προσέγγιση. Ε, θα ήθελα να δω τα πράγματα σε... Ε, από τρεις απόψεις. Πρώτα-πρώτα για το ταμείο που θα δημιουργηθεί. Οι χώρες ας πούμε όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και τα που, είναι, που έχουν μεγαλύτερη, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κρίση και μπορεί να γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπιών επιθέσεων ε, θα πρέπει οι χώρες αυτές κάπου να μπορέσουν να υποφεληθούν από το ταμείο αυτό η Ισπανία βεβαίως η Ισπανία βεβαίως ήταν ο καλός ο μαθητής ε, και έχει κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν ξέρουμε όμως αν θα πρέπει να μπει απαραίτητος του ε, Ταμείο του Χρέους ή όχι από εκεί και πέρα για το 60% του χώριου προϊόντος τα μπλε και τα κόκκινα ομόλογα Ιταλία η Ιταλία ε, είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία. Ε, λέμε εδώ 25 χρόνια. Ε, έχω την εντύπωση ότι πρώτα πρώτα να δούμε ότι στην Ιταλία δόθηκαν ουσιαστικά τρία χρόνια για να κάνει ορισμένες αλλαγές. Δεν ξέρω κατά πώς θα τα καταφέρει ο κ. Μόντι, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ μιλάμε για διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Από εκεί και πέρα ε, υπάρχουν και άλλες πτυχές που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, να ξεχνούμε την ανάπτυξη, την απασχόληση, καταπολέμηση της ανεργίας ε, όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα ξεχνούμε υπάρχουν πάρα πολλά με στο πλαίσιο το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τώρα Μάρκους, ευχαριστώ πολύ Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα να πω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. τι θα πει αυτό. Θα πει ότι οτιδήποτε σχετίζεται με ενδεχόμενη τροποποίηση των συνθήκων ε, είναι μη ρεαλιστικό. Ε, δεν μπορούμε να το αναλάβουμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή όποιος πιστεύει ότι μπορούμε να κάνουμε από τη μια στιγμή στην άλλη 27 ε, χώρες τροποποίηση των ε, συνθήκων για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτά πατάτε ε, δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι ουτοπικό να ξεκινούμε από την υπόθεση ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι παραμένουν οι συνθήκες και πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Για να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ποια είναι η αιτία της υπερβολικής ανάληψης χρέους από ορισμένε χώρες. Οι χώρες αυτές ε, ιστορικά τι επιτόκια είχαν. Ε, άμα η, τα επιτόκια με τα οποία δανειζόντουσαν οι χώρες αυτές ήταν ιστορικά χαμηλά τότε γι' αυτό δανείζονταν, δανείστηκαν υπερβολικά οι χώρες δείτε τι γίνεται με τις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και θα το δείτε εγώ ε, εδώ λοιπόν θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και να δούμε και τη λύση την οποία προτείνουμε να μην προτείνουμε, να προτείνουμε πράγματι φάρμακο και όχι ε, ναρκωτικό για την εξηγένση των χωρών αυτών ε, που αποβλακώνει αν θέλετε περισσότερο τις χώρες αυτές διότι και αν τα σκεφτούμε αυτά καλά θα δούμε ότι ναι μεν η κοινή εξόφληση του χρέους δεν, η από κοινού εξόφληση του χρέους δεν είναι κακό πράγμα αλλά η από κοινού πλήρης εξόφληση του χρέους κατά 100% όπως προτείνεται εδώ είναι αυτό το ναρκωτικό που έλεγα και το θεωρώ πάρα πολύ κακό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε τη τη βιωσιμότητα αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος θα πρέπει να βρούμε διαφορετικές λύσεις. Λοιπόν, τώρα για το κείμενο της Κομισιόν και τις τρεις επιλογές που προτείνει είμαι πολύ διστακτικός. Ε, έχω προτείνει εγώ κάποιες αλλαγές μέσω των τροπολογιών μου ε, και θα επιμείνω σε αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank και εγώ ευχαριστώ. Αστρίτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι μεγάλο μέρος των διακοπών μου ε, με απασχόλησε με την ανάλυση των 250 τροπολογιών ε, της εκθέσεως ε, της ε, συναδέλφου Γκολάρ. Και με τον τρόπο αυτό διαπίστωσα την ε, δυσκολία που αντιμετωπίζει συνάδελφος έτσι ώστε να καταφέρει να βρει μια λογική συμφωνία μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ε, μεγάλων αποκλήσεων που παρουσιάζει η Επιτροπή μας. Αυτό που θεωρώ εγώ ουσιαστικό και μια και οπωσδήποτε κατά την άποψή μου θα πρέπει να οδηγηθούμε προς ε, μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Αυτό που είναι λοιπόν ουσιώδες είναι ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε και σε μεγαλύτερη πειθαρχία. Και το ένα θα πρέπει να ακολουθεί το άλλο. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο αλληλεγγύης που είναι τα ευρωομόλογα. Ε, δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να ανοίξουμε εμείς πρώτοι και το δρόμο της πειθαρχία. Κατά την άποψή μου προχωράμε με πολύ μικρά βήματα ε, και τα κείμενα που ψηφίσαμε και όσον αφορά τις ε, προτάσεις για το παρόν και για το μέλλον κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε ένα τόσο περίπλεκο σύστημα το οποίο ε, ε, δεν θα οδηγήσει τελικά σε καλά αποτελέσματα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη μονάχα ένας εξάντε έλεγχος των, εκ των προτέρων, δηλαδή έλεγχος των εθνικών προϋπολογισμών θα μπορέσει να οδηγήσει στις πραγματικές διαρροτικές αλλαγές τις οποίες χρειάζεται ο επιγόντος η Ευρωζώνη. Όσον αφορά τώρα ε, τον τρόπο εφαρμογής. Ε, φυσικά όλοι οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί ε, και το, η πόρτα του Συμβουλίου θα πρέπει να ανοιχτεί για νέες διαπραγματεύσεις. Βεβαίως φαίνεται περίπλοκο ακόμα και το θέμα της ανάληψης ευθύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, που δεν στηρίζεται σε πολύ έτσι, σταθερούς ώμους αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, έτοιμες λύσεις δεν υπάρχουν και το βέβαιο είναι ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο ε, να πει κάτι παραπάνω σε μια έκθεση πρωτοβουλίας από το απλώς να δηλώσει ότι χρειαζόμαστε ευρωομόλογα, γιατί έτσι δεν θα μας ακούσει κανένας. Ε, βλέπω ότι έγιναν ενδιαφέρουσες προτάσεις από τον ε, Ισπανό Υπουργό ε, για δράση σε τρεις φάσεις που νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να τις ακούσουμε. Εγώ επιμένω στο ότι οποιαδήποτε αποφασιστική πρόοδος προς την αμοιοβιοποίηση του χρέους θα πρέπει να βασίζεται σε εξάντε έλεγχο των προϋπολογισμών ε, και βεβαίως θα πρέπει να ακολουθηθεί ε, και από δικαίωμα βέτο αρνησικυρίας από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε εθνικό προϋπολογισμό ο οποίος δεν σέβεται τις από κοινού σε ε, υποχρεώσεις και ευθύνες. Πέραν τούτου δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο να βρούμε ε, κοινό τόπο συνεννόησης εάν ε, δεν μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια κοινή οδό αλληλεγγύης αλλά και πειθαρχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των συντηρητικών πρέπει να πω ότι ε, δεν είμαι ε, υπεύθυνο και σκιώδης ε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο συνάδελφος ε, ε, βρίσκεται στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, οπότε δεν είναι εδώ. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορέσει λοιπόν να πάρει τον λόγο εξ των συντηρητικών. Έχει υποβάλει βέβαια πολλέ τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες γενική εφήσεως παρατηρήσεις επί του θέματο αυτού το οποίο βεβαίως θεωρούμε ουσιώδους και μεγάλης σημασίας, όχι μόνο όσον αφορά τον τύπο αλλά και κυρίως όσον αφορά το περιεχόμενο. Επί τη βάση λοιπόν των όσων ελέγχθησαν μέχρι τώρα από τους προηγούμενους συναδέλφους θα συμφωνήσω ότι χρειαζόμαστε βεβαίως μια γρήγορη και έγκαιρη αντίδραση. Όμως το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Η ταχύτητα είναι πάντα ο καλύτερος σύμβουλος. Γιατί ε, ε, αν μιλάμε για ομόλογα, για μένα το κυριότερο ζήτημα πρέπει να είναι γενικότερο. Δηλαδή, σε τι ανταποκρίνονται τα ευρωομόλογα στα βραχυπρόθεσμα προβλήματα ή αντιμετωπίζουν ε, τις ανισορροπίες οι οποίες εδώ και δεκαετίες υπάρχουν στην Ευρώπη, απλώς εμφανίστηκαν στην πλήρη τους μορφή τώρα. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, βρούμε ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο και θα μπορεί βεβαίως να, αντιμετωπίσει, ε, να αντιμετωπίσουν προβλήματα μεσοπρόθεσμα. Αν όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε βρα, συγγνώμη, μακροπρόθεσμα προβλήματα, πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι πλέον. και αν ε, τα κράτη-μέλη μεμονωμένα κάνουν διαφορετικές ε, ε, τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σε κάποια καλά αποτελέσματα, αυτό είναι καλό. Σε αντίθετη περίπτωση όμως θα επιταχυνθεί ο δημοσιονομικός κίνδυνος. Δεύτερον, και εδώ πρόκειται για τροπολογία του συναδέλφου Ήπινγκ, με κανένα τρόπο τα ομόλογα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αποτελέσουν εργαλείο αύξησης ε, της ε, ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ε, είναι ψεύδος εάν πει κανείς κάτι τέτοιο. Τρίτον, τα ευρωομόλογα μπορούν να λύσουν κάποια προβλήματα, ε, αλλά αναφέρονται σε ένα οικονομικό και κοινωνικό χώρο που δεν είναι ομοιογενής, είναι εξαιρετικά ετερογενής και επομένως θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αρνητικά και όχι θετικά. Ε, φτάνω και σε κάτι άλλο, του οποίου είμαι εγώ συγγραφέας, ε, αναφέρομαι εδώ στην πολιτική διάσταση. Πιστεύω ότι η χρήση των ευρωομολόγων χρειάζεται, απαιτεί τροποποίηση των συνθήκων και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Σκεφτείτε λίγο τι έγινε στις κάτω χώρες και στην ε, Γαλλία, ε, στην ε, ψηφοφορία, στο δημοψήφισμα μάλλον, για την για το, για το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Επομένως, σκεφτείτε λίγο, αναλογιστείτε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις ε, και σε αυτή την περίπτωση. Ε, επομένως, εάν αμφισβητηθεί ο ευρωπαϊκός χώρος, αυτό θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα άσχημα αποτελέσματα όσον αφορά την ευρωπαϊκή συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ε, να σας υπενθυμίσω ότι ενδεχομένως ε, ε, θα χρειαστεί να σταματήσουμε πέντε λεπτάκια πιο πριν ε, από τις και μισή για να ετοιμάσουμε την αίθουσα για το κεκλεισμένο των θυρών με τον κύριο Ντράγκη. Λοιπόν, θα κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, το πρόβλημα με το άχθος των επιτοκίων ε, για τις χώρες είναι υπαρκτό. Και επομένως, ε, ακόμα και αν ορισμένοι προσπαθούν να ε, το καταδικάσουν αυτό, η αμοιβαιοποίηση του χρέους ήδη συμβαίνει από την αρχή του ο, ο, του, της κρίσης. Ε, κατά 2,6 έχει αυξηθεί ο ισολογισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, και ε, στην ουσία τώρα χάνουμε στην ουσία το, το, κρίσιμο σημείο, δηλαδή ότι ήδη είτε το θέλουμε είτε όχι, το παραδεχόμαστε είτε όχι, οδηγούμαστε στην αμοιβαιοποίηση του χρέους και επομένως δίνουμε όλο και περισσότερα χρήματα στο οικονομικό σύστημα της Ευρώπης χωρίς καμία δημοκρατική διαφάνεια ή λογοδοσία η ε, ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και θα πρέπει να κάνει μια ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Και εδώ επομένως θα πρέπει να κάνει νομισματική πολιτική και όχι οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική θα πρέπει να υφίσταται την δημοκρατική διαδικασία και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ε, αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα τώρα. Και επομένω ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε μεμονωμένε αποφάσει για θέματα τα οποία είναι πολύ ε, πολιτικά. Όσον αφορά δε το Ταμείο Εξόφλησης του Χρέους, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και άλλωστε υπάρχει και μία πρόταση των σοφών της ε, Γερμανίας. Ε, να ε, δοθεί δηλαδή κάποιο είδους ασφάλεια ή διασφάλιση από τις χώρες οι οποίες θα μπουν στο σύστημα αυτό. Γιατί τούτη τη στιγμή αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι μια πρόταση η οποία ενδεχομένως θα στηριχτεί πολιτικά. Δεν σημαίνει τίποτα το να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει ό,τι θέλει να ασκήσει πολιτική χωρίς να έχει όμως τον πολιτικό έλεγχο έλεγχο. Και εκπλήσωμαι, γιατί πολύ συχνά αυτοί που είναι κατά των ευρωομολόγων, κατά του ε, Ταμείου Εξόφλησης ε, Χρέους, κριτικάρουν την, ε, είναι αυτοί που κριτικάρουν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα στις χώρες τους ε, και στην ουσία χάνεται ε, η πολιτική στήριξη προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, πράγμα που δεν πρέπει να συμβεί. Και όσον αφορά τώρα το θέμα των ε, μακροπρόθεσμων ε, ε, ευρωομολόγων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε για την μακροπρόθεσμη ατζέντα, γιατί ενδεχομένως θα είναι καλύτερα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, έχει ψηφίσει και το Κοινοβούλιο και πριν από την κρίση όσον αφορά τα ευρωομόλογα και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σε βράχη πρόθεσμη βάση τα ευρωομόλογα δεν μπορεί να μας βοηθήσουν, αν δεν υπάρχει κατάλληλη αιρεσιμότητα κτλ. Όμως όμως εάν θέλουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά όλα τα εργαλεία για την αμοιβαιοποίηση θα πρέπει ε, να είμαστε πρώτον έντιμοι στη συζήτηση που κάνουμε και δεύτερον να στηρίξουμε οπωσδήποτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. η σοφή. Ευχαριστώ Σάρον. Θα προσπαθήσω και σύντομη ναι, αλλά και να απαντήσω σε όλους. Θέλω να απαντήσω πρώτα στο ρόλο. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας αυτή και εγώ με τους Σκιώδη συζήτησα πρώτα κατά πολύ και την είδαμε σαν ε, μία παρουσίαση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Δεν μπορούμε βέβαια να τα συμπεριλάβουμε όλα, αλλά προκειμένου να ξεκινήσει μια δημόσια, ανοιχτή και δημοκρατική συζήτηση πάνω στις διάφορες εναλλακτικέ. Κάτι πολύ σημαντικό το είπε και ο Φιλίπ Λαμπέρ, αλλά το λέω και προς τον κύριο Φέρμπερ, είναι το εξή. Στη συνθήκη, ή μάλλον στην έκθεση, υπάρχει ιδέα του χάρτη πορείας. Γιατί, Γιατί εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένη ότι δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τη συνθήκη, παραβιάζοντας δηλαδή τη συνθήκη. Αν διαβάσετε λοιπόν την έκθεση προσεκτικά, θα δείτε ότι η έκθεση αυτή, σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται σε πολλές χώρες, λαμβάνει υπόψη τα νομικά επιχειρήματα τα οποία ανέφερε. Εκεί που έχετε δίκιο είναι όταν λέτε ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε μια συζήτηση, συζήτηση που να κρύβει κάποια πράγματα. Τη συνθήκη θέλουμε φυσικά να την τηρούμε και να τη σεβόμαστε, αλλά αν δεν πάρουμε καμία πολιτική απόφαση, οι συνθήκες θα γίνουν από το οποίο κρυβόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Όλες οι μεταφορές που γίνονται μέσω του μηχανισμού Target 2 της Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Απ' τη μια υπάρχει αυτή η παρθενιά ας πούμε των συνθήκων και απ' την άλλη υπάρχουν αυτοί που θέλουν να την παραβιάσουν. Λοιπόν, ειλικρινά, το να λέμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, όχι, πρέπει να λέμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι οι ορισμένες οικονομίες ανησυχούν για την σταθερότητα μακροπρόθεσμα της ζώνης του ευρώ. Δεν λέω εγώ ποια είναι η καλύτερη λύση. Λέω όμως ότι υπάρχουν αναλλακτικέ και πρέπει να καταλήξουμε κάπου. Η πραγματικότητα μας έχει ξεπεράσει, πρέπει να ξέρετε. Για να απαντήσω τώρα στην Άστρι Λούλινγκ. Μα δεν είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης αυτό που προτείνω εγώ. Αντίθετα, πώς μπορούμε με φύ τρόπο να έχουμε πειθαρχία έτσι ώστε να μην χρειάζεται αλληλεγγύη που να μην την έχουμε προβλέψει. Γιατί σήμερα αρνούμαστε ε, κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν την πειθαρχία. Και επειδή ήμουν εισηγήτρια για τη δέσμη των 6 μέτρων και με τη γαλλική κυβέρνηση την τότε είχα αγωνιστεί για να ενισχυθεί η πειθαρχία. Δεν είναι θέμα επιλογής πειθαρχία ή όχι πειθαρχία. Όχι. Είναι πώς θα έχουμε πειθαρχία με φύ τρόπο, με μηχανισμό δηλαδή να ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες εκείνες οι οποίες βρίσκονται στην παγίδα μέσα. Χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε καθόλου την πειθαρχία. Κάθε άλλο. Τώρα για τον εξάντε έλεγχο των προπολογισμών νομίζω ότι λίγο-λίγο τα καταφέρνουμε. Και με την δέσμη των 6 μέτρων και με το ευρωπαϊκό εξάμενο, με όλα αυτά που πρέπει τα κράτη-μέλη να δίνουν πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν εγκρίνει τον προπολογισμό τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμησε ότι σκοπός της είναι να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα. Τέλος, θα δούμε βέβαια λεπτομερώς όλες τις τροπολογίες και με τους σκιώδες και με την ομάδα μου και όπως λέει και ο Διέγο, ο Εντουαρ δεν είναι εδώ, αλλά να ξέρετε ότι οι σκιώδεις βοηθούν πάρα πολύ για να έχουμε μια κοινή βάση. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Δεν πρόκειται τώρα να αποφασίσουμε οριστικά εντοπίζουμε τις λύσεις που υπάρχουν, που είναι καλύτερες από κάποιες άλλες. Και ακούστηκαν και κάποιες νέες ιδέες. Ο Ρωμάνο Πράντη έγραψε ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα, ο τέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μιλούσε για εγγύσεις σαν και αυτές που θέλουμε και εμείς με το Ταμείο Εξόφλησης του Χρέους, ώστε κοινή ευθύνη να μην βαραίνει περισσότερο κάποιες χώρες από ό,τι κάποιες άλλες. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και τεχνικά μέσα που μπορούν να βοηθήσουν. Πάντως εδώ το θέμα είναι να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά και όχι που ο καθένα να την κάνει για να πάει μετά στην εκλογική του περιφέρεια και να πει «Α, εγώ πέρασα το μήνυμα που θέλατε». Όχι. Είτε πρόκειται για ε, να πούνε ότι α, τηρούμε τους κανόνες που τελικά δεν τους τηρούμε ή να πούμε ότι α, εμείς κάνουμε προσπάθειες, όχι όλοι κάνουμε προσπάθειες. όσες ε, τροπολογίες έχουν επικοδομητικό πνεύμα θα τις ε, στηρίξω και όχι τις άλλες. Μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε τη σταθερότητα ολόκληρη της Ευρωζώνης που έχει να κάνει με όλους τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. θα ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε τον Οκτώβριο να πάει η έκθεση αυτή στην Ολομέλη. Εννοείται ότι μένει πολλή δουλειά να γίνει με τις τροπολογίες μέχρι τότε. Συνεπώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν σύντομοι. Τώρα, παρακαλώ, όσοι δεν προβλέπεστε για την κεκλεισμένον των ε, θυρών συνεδρίαση να φύγετε για να υποδεχτούμε εδώ τον κύριο Τράκη και τον κύριο Μπαρνιέ. Και μετά για τον προπολογισμό και τις ψηφοφορίες μπορείτε να επανέλθετε. Μόνο λοιπόν, το λέω και το επαναλαμβάνω, οι ευρωβουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να μείνουν εδώ. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή πρέπει να φύγουν, τα Εθνικά Κοινοβούλια να βγούνε, ούτε οι λόμπις δεν επιτρέπεται να μείνουν εδώ, ούτε εκπρόσωποι του τύπου. Αν υπάρχει κανένας που βλέπετε περίεργο σαν κατάσκοπο, πείτε το μας να τον πετάξουμε έξω. Ο λόγος είναι ότι προβλέπονται πειθαρχικέ ε, διαδικασίες και δεν μπορώ λοιπόν να επιτρέψω να μείνουν εδώ άτομα τα οποία δεν είναι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό παρακαλώ να καταλήψετε την αίθουσα. And I also have Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εννοείται δεν μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίε ούτε και να ηχογραφήσετε τίποτα. Δεν χρειάζεται να σας το υπενθυμίσω αυτό. Απαγορεύεται η ηχογράφηση, απαγορεύονται οι φωτογραφίες. Και φροντίστε ε, το web streaming να έχει κλείσει, να μην περνάει στο διαδίκτυο η συνεδρία σε αυτή πια.